πράγματα και δείχνοντα αλληλεγγύη και για τρίτες χώρε. Αυτές ήταν οι προτεραιότητές σα Στη θεωρία ήρθε η ώρα όμω να περάσουμε από τα λόγια στα έργα και να τις συγκεκριμενοποιήσουμε. Ο κύριος Μάγερ για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχά, ε, καλώ επιστρέψατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κύριε Πρωθυπουργέ. Στην αρχή τη παρέμβασή σα αναφερθήκατε σε τρία ζητήματα. Το πρώτο ήταν το πολιτέ νομοσυνομικό πλαίσιο, το δεύτερο ήταν το Brexit και τέλο αναφερθήκατε στη διεύρυνση. Θεωρώ πραγματικά ότι πολύ σωστά επιλέξετε τα ζητήματα αυτά ω τα πιο σημαντικά και τα πιο επίγοντα. Πιστεύω ότι όντω θα πρέπει να δημιουργήσουμε την απαραίτητη σταθερότητα όσον αφορά τη χρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερον, θα πρέπει να χάσουμε την ευκαιρία να διαπραγματευτούμε μια καλή συμφωνία με το Μένο Βασίλειο και τρίτον, α αποφύγουμε οποιαδήποτε αποσταθεροποίηση τη περιοχή τη περιοχή των Βαλκανίων. Υπάρχει όμω και ένα ακόμα πιο σημαντικό ζήτημα. Η πρόεδρο Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η κυρία Φοντελάν, αναφέρθηκε στην, στον ενθουσιασμό τη Προεδρία σα και αναφέρθηκε επίση και στην εμπειρία σα. Το είπε αυτό και ο κύριο Βέμπερ. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να έχουμε μια πιο ισχυρή συνεργασία μεταξύ ημών και να καταφέρουμε τελικά να κάνουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση πιο ενωμένη, πιο συλλογική. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία. Κυρία Φαγιόν, τώρα έχει το λόγο και ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Πρωθυπουργέ, πραγματικά μπροστά σας έχετε κάποιες πολύ σημαντικές προκλήσεις. Δεν μπορώ λοιπόν παρά να υποστηρίξω τις προτεραιότητές σας. Ωστόσο, νομίζω ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε στο ζήτημα του κράτους δικαίου. Νομίζω ότι ε, θα πρέπει ε, πάση θυσία να καταπολεμήσουμε τη ρητορική μίσου και να χειριστούμε αποτελεσματικά τη μετανάστευση. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά και για το μέλλον του χώρου Σέγγεν. Είναι προ το δικό μα συμφέρον να ενταχθεί το συντομότερο δυνατό η Κροατία στο χώρο Σέγγεν. Πριν γίνει όμω αυτό, θα πρέπει να εμφυσίσουμε νέα εμπιστοσύνη στους Ευρωπαίους πολίτες, θα πρέπει να προστατεύσουμε τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει ο χώρος Σέγγεν να γίνει πιο αποτελεσματικός. Συμφωνώ ότι θα πρέπει να προωθήσουμε την ευρωπαϊκή προοπτική των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων και ήδη πιστεύω ότι από το Μάρτιο θα πρέπει να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις με την Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία. Οι ε, δυο μας χώρες, η Κροατία και η Σλοβενία, θα πρέπει να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να ενισχύσουν τη μεταξύ ημών συνεργασία. Σας ευχαριστούμε ο κύριος Κούμπιλους. Έχει το λόγο για ένα λεπτό. Κύριε Πρωθυπουργέ, Είμαι από τη Λιθουανία και χαίρομαι ιδιαίτερα που μπορώ να σας συγχαρώ, κύριε Πρωθυπουργέ, και εσάς αλλά και ε, το λαό της χώρας σας για την πρώτη Προεδρία που αναλαμβάνετε. Κάτι πολύ σημαντικό, λόγω και της υψηλής ε, συμβολικότητας ε, της Προεδρίας σας, 25 ε, χρόνια μετά το τέλος του πολέμου της ανεξαρτησίας ηγείται όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Κροατία. Είναι το πλέον πιστικό παράδειγμα του πώς μπορεί η Ευρώπη να φέρει την ευημερία μέσω της διεύρυνσης στις γειτονικέ χώρες. Είναι θαύμα και πολύ σωστά είπε ότι η επαγγελία ε, για την διεύρυνση είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κίνητρο για τις μεταρρυθμίσεις χώρες ε, και ε, είναι πολύ μεγάλη έμπνευση για τις άλλες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων η Κροατία. Η και για τις χώρες της ε, Ανατολικής Γειτονίας είναι έμπνευση και ελπίζω όταν γίνει η σχετική διάσκεψη να χαρακτηρίζεται από μεγάλη φιλοδοξία και να εμπνεύσει την περιφερειακή στρατηγική για την επόμενη δεκαετία. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία κύριε Πρωθυπουργέ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Λαλίκ. Λαλίκ. Ένα λεπτό. Αγαπητέ Πρωθυπουργέ, κυρίες Πρόεδροι, το οικονομικό μοντέλο σήμερα πνέει τα λίστια. Αν καταφέραμε μεν να βγάλουμε δισεκατομμύρια από την ε, φτώχεια, ε, αυτό οδήγησε σε μια δραματική κατάσταση σήμερα. Δεν μπορούμε να βελτιώσουμε ε, το περιβάλλον και δεν μπορούμε να βελτιώσουμε και τις κοινωνικές συνθήκες στην Ήπειρο. Το οικονομικό μοντέλο δεν μπορούμε να το μεταρρυθμίσουμε. Έχουμε αυτή την ψύχωση με το ΑΕΠ, κάτι παράλογο αν δει κανεί ε, και τους δείκτες ε, που δεν μπορούν να μας πούν τίποτα για τις ανισότητες, για την κατάσταση του περιβάλλοντος, για τη φτώχεια. Επιλέξατε η Προεδρία σας να είναι για μια ισχυρή Ευρώπη που θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της. Και η μεγαλύτερη πρόκληση, κατά τη δική μου άποψη, που έχετε να αντιμετωπίσετε είναι να αλλάξουν οι δείκτες ε, που καθορίζουν τον πλούτο. Να αλλάξει, αν θέλετε, ε, εντό αγωγικών ε, το θεσμικό λογισμικό. Εμείς σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία και βασιζόμαστε σε εσά. Σας ευχαριστώ. Για ένα λεπτό, το λόγο έχει η κυρία Τόμτς. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Πρωθυπουργέ Πλένκοβιτς, αγαπητέ Αντρέη, εγώ έχω εμπειρία από την άσκηση Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέρω πόσο δύσκολο είναι και τι σημαίνει αυτό και σας εύχομαι καλή επιτυχία. Από τις προτεραιότητες σας διάλεξα την ανάγκη ανάπτυξη. Θέλουμε μια ισορροπημένη ανάπτυξη και η συνοχή είναι απαραίτητη όχι μόνο για τις χώρες δικαιούχου, αλλά για όλα τα κράτη-μέλη. Αν όλα τα κράτη ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά του, θα ενισχυθεί η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, θα ήθελα να αναφερθώ στις προκλήσει της δημογραφίας. Είναι όλο και πιο σημαντικό το δημογραφικό πρόβλημα και κυρίως ε, στη δυτική περιοχή. Ας μην ξεχνούμε τη γύρεση του πληθυσμού, την υπογεννητικότητα και το γεγονός ότι οι νέοι μας αποδημούν στο εξωτερικό. Και όλα αυτά τα θέματα είναι αλληλένδετα. Ε, και κυρία Επίτροπε Σουίτσα, πιστεύω ότι θα δραστηριοποιηθείτε ιδιαίτερα και σας εύχομαι καλή επιτυχία. Ευχαριστώ για ένα λεπτό, ο κύριος Χάισερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε της Κρατικής Κυβέρνησης, μια ισχυρή Ευρώπη σε ένα κόσμο γεμάτο προκλήσεις είναι πολύ εύστοχο σύνθημα και σλόγγαν της Προεδρίας σας, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ισχύ. Θα πρέπει λοιπόν να τη χρησιμοποιήσει και να την αξιοποιήσει αποτελεσματικά. Θα πρέπει για να γίνουμε οικονομική υπερδύναμη να αξιοποιήσουμε αυτή την έλξη που ασκούμε σε άλλες χώρες. Και θα πρέπει να είμαστε ανοιχτοί, ε, αλλά ταυτόχρονα να εκφέρουμε τις άποψή μας με ενιαία φωνή, να υπάρχει ομοφωνία και σύμπνοια. Έχουμε πολλές προκλήσεις και θα χρειαστεί χρηματοδότηση πολλών πολιτικών. Αυτή ίσως θα είναι και η πιο σημαντική πρόκλησή σας. Θα πρέπει να μεριμνήσουμε όλοι ώστε ε, να συμβιβάσουμε τα συμφέροντα των αμυγών συνεισφορέων με εκείνα των δικαιούχων που συνεισφέρουν λιγότερο και εξαρτώνται περισσότερο από τα διαρθρωτικά ταμεία όπως ε, η Κροατία και η Σλοβακία η χώρα μου. Ο κύριος Χριστοφόρ. Αγαπητέ φίλε Πρωθυπουργέ της Κροατίας, θα ήθελα πραγματικά να σας ευχηθώ από καρδιά καλή επιτυχία και είμαι πεπισμένος γνωρίζοντας τις ικανότητες και τις δυνατότητές σας ότι μπορείτε να ισχυροποιήσετε την ευρωπαϊκή ένωση και να δημιουργήσετε μια πιο αναβαθμισμένη εικόνα στους ευρωπαίους πολίτες. για να καταστεί τούτο δυνατό όμως χρειάζεται ισχυρή οικονομία και απαιτείται ένα ισχυρό πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο με την αύξηση της συνεισφοράς των χωρών μελών απαιτείται ισχυρή άμυνα και ασφάλεια και συμφωνώ μαζί σα ότι δεν μπορεί να υπάρξει ευρωπαϊκή ένωση χωρί να διασφαλίσουμε τα σύνορά μα και απαιτείται αυστηρή προσήλωση σε αρχέ και αξίε όμω η ευρωπαϊκή ένωση δεν μπορεί να καθίσταται παρατηρητή είτε στη λιβύη είτε στη συρία και δεν μπορεί να αφήνει και να ανέχεται χώρε όπω την τουρκία ουσιαστικά να δημιουργούν αποσταθεροποίηση στην περιοχή αλλά και να απειλούν χώρε μέλη τη ευρωπαϊκή ένωση όπω η κύπρο και η ελλάδα. συμφωνώ απόλυτα με την αγαπητή πρόεδρο τη ευρωπαϊκή επιτροπή ότι όπου υπάρχει ενότητα υπάρχει πραγματικά ελευθερία. θα προσθέσω όπου υπάρχει αλληλεγγύη υπάρχει ενότητα υπάρχει και ελευθερία και αυτή τη στιγμή δύο χώρε μέλη τη ευρωπαϊκή ένωση αγαπητή κυρία πρόεδρε η κύπρος και η ελλάδα ζητούν έμπρακτα την αλληλεγγύη σας απέναντι σε μια χώρα τρομοκράτη όπως είναι η τουρκία που δημιουργεί αστάθεια στην περιοχή. ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Μωρέτη. Έχει τώρα το λόγο για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε Πλένκοβιτς, ε, κυρία Φοντελάιεν, αγαπητοί συνάδελφοι. Κλειδονίζεται ο κόσμος γύρω μας από τον πόλεμο και τις εντάσεις και παρόλα αυτά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν συμμετέχει καθόλου, είναι ουραγός δεν έχουμε το θάρρος να πάρουμε συγκεκριμένε θαραλέες αποφάσεις. Είμαι πεπισμένη πάντως ότι έχοντας μια γυναίκα πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπως η Ούρσουλα Φοντελάιεν μπορεί πραγματικά να αλλάξει τα δεδομένα. Δύο σημαντικές επιλογές θεωρώ ότι θα είναι καθοριστικές στο μέλλον. Όσον αφορά το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο καταρχάς. Επ' αυτού θα πρέπει πραγματικά να τα αποκρίνετε στις προκλήσεις και η πρόταση της φιλανδική προεδρία θεωρώ ότι υπολείπεται του επαρκούς επίπεδου χρηματοδότησης και σε καμία περίπτωση δεν μας επιτρέπει να ελοποιήσουμε το πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο εμεί εγκρίναμε ω Ευρωβουλευτέ. Επίση, δεν θα μπορέσουμε να δώσουμε τη σύμφωνη γνώμη μα για το πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο αν δεν αλλάξει το σύστημα ιδίων πόρων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίση, η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία θα πρέπει να αποτελέσει επανάσταση, όχι μόνο οικονομική, αλλά και κοινωνική και οικολογική. Θα πρέπει πραγματικά να δημιουργήσει βιωσιμότητα χωρί να αφήνει πίσω κανέναν. Ζητώ λοιπόν από την Κροατική Προεδρία να επιμείνει, διακόπτη η Πρόεδρο. Σας ζητώ συγγνώμη, αλλά εξέπνευσε ο χρόνος που είχατε. Η κυρία... Γκλάβα και επόμενη ομιλήτρια για ένα λεπτό επίσης. Ευχαριστώ. Κύριε Πρωθυπουργέ της Κροατίας, η Κροατία με την ιστορία της έδειξε ότι δεν φοβάται τις προκλήσεις και η Κροατική Προεδρία θα είναι ευκαιρία να δείξει ε, ευθύνη απέναντι στους πολίτες πρώτα απ' όλα και υπευθυνότητα. Θέλουμε μια Ευρώπη ε, που αναπτύσσεται, όπου μεγάλοι και μικροί, φτωχοί και εύποροι έχουν ισότιμες ε, και παρόμοιες ευκαιρίες και θα πρέπει να ε, γίνει μια κρυβοδίκη κατανομή των ε, οικονομικών μας πόρων στα πλαίσια του νέου πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου. Πρώτα απ' όλα όμως θα πρέπει να επαναφέρουμε και να αποκαταστήσουμε την ε, εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων πολιτών στη γυραιά Ήπειρο, που θα πρέπει να είναι διορθωτικός ο χαρακτήρας της και να ανταποκρίνεται και να αντιμετωπίζει τις νέες προκλήσεις. Γιατί ε, όσοι δεν γνωρίζουν την Κροατία δεν, γνωρίζουν, δεν γνωρίζει πώς η οικονομική της ε, ανάπτυξη είναι σημαντικό θετικό μήνυμα. Είμαστε έτοιμοι για τις ε, προκλήσεις, θα διαρωτούνται πολύ Σας πληροφορώ ότι είμαστε πανέτοιμοι και θα δείξουμε ότι είμαστε στο ύψος των περιστάσεων. Σας ευχαριστώ. Για ένα λεπτό κύριε Γιούρη, περνάμε στη διαδικασία του Catch the Eye. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρωθυπουργέ. Να συγχαρώ, να συγχαρώ μάλλον για το πρόγραμμα που μας παρουσιάσετε τη Κροατική Προεδρίας. θα πρέπει να συνεχιστεί προφανώ η συζήτηση που γίνεται τελευταία χρόνια για το κράτο δικαίου. Νομίζω δεν θα πρέπει να απομονώνουμε συγκεκριμένες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης το κράτος δικαίου δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σαν παιχνίδι, σαν εργαλείο, προκειμένου να διευθετούμε τις διαφορές που έχουμε με συγκεκριμένε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανταυτού νομίζω ότι θα πρέπει όλες οι χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης ισότιμα να αξιολογούνται για το πώς εφαρμόζουν το κράτος δικαίου. Να ισχύουν για όλες τις χώρες οι ίδιοι κανόνες και τα ίδια κριτήρια. Και ας μην συγχαίουμε αυτή τη στιγμή τα εσωτερικά καθαρά ζητήματα που δεν έχουν να κάνουν με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τα ευρωπαϊκά ζητήματα. Σας παρακαλώ πολύ λοιπόν, ας μην είμαστε εμείς ε, οι εξωτερικοί κριτές για καθαρά εσωτερικά ζητήματα. Αυτή τη στιγμή διακόπτη η Πρόεδρος, ολοκληρώθηκε ο χρόνος αγόρευσης. Η κυρία Μάρκη έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον Κροάτη Πρωθυπουργό να ευχαριστήσω, επαναλαμβάνω, τον Κροάτη Πρωθυπουργό για την παρουσίαση των, προτε... των προτεραιοτήτων της κρατικής προεδρίας, μεταξύ αυτών και της προτεραιότητας για την διεκπαιρέωση των συζητήσεων και την υιοθέτηση του νέου ΠΔΠ πολιτούς δημοσιονομικού πλαισίου. Επίσης, με τεράστια ικανοποίηση, άκουσα να λέτε πόσο σημαντικό είναι να διαφυλάξουμε στο νέο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο την αξία της πολιτικής συνοχής και της κοινή γεωργικής πολιτικής έχουμε επιτάπητος μία πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, λέει ότι 7,5 δισεκατομμύρια νοπό χρήμα θα, θα ε, εφοδιάσουν το νέο Ταμείο Δικής Μετάβασης. Επίσης, ε, είχαμε τις προτεραιότητες προηγούμενης Προεδρίας της Φιλανδικής ε, και θα ήθελα να ε, ρωτήσω ποιες είναι οι δικές σας απόψεις σχέση με τις προηγούμενες ε, προτεραιότητες, προηγούμενες Σας ευχαριστώ κυρία Γιώβερα. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πλένκοβιτσα, σα ευχαριστούμε που μα παρουσιάσατε τι προτεραιότητε τη κροατική Προεδρίας. Μια Προεδρία που αναλαμβάνεται σε ταραχώδει καιρού, όπου αναμένουμε πολλέ αλλαγέ. και είτε το θέλουμε είτε όχι υπάρχουν ζητήματα όπω ο προπολισμός του μέλλον τη Ευρώπη, το Brexit, περιβαλλοντική νομοθεσία που θα είναι στο προσκήνιο. Κάποια από αυτά τα θέματα τα έχετε επιλέξει και εσεί. Μεταξύ αυτών θα ήθελα να μιλήσω για τι δημογραφικέ αλλαγέ, τη διεύρυνση προ τα Δυτικά Βαλκάνια και το σεβασμό των θεμελιωδών των αξιών τη Ένωση, όπω είναι το κράτο δικαίου. Η δική σα χώρα, η κροατική δική μου χώρα, η Σλοβενία, είναι γειτονικέ χώρε. και θεωρώ ότι θα έχουμε πολύ καλή συνεργασία αυτό το εξάμεινο και ακριβώ λόγω αυτού βασίζομαι και σε εσά, κύριε Πλένκοβιτ, να κάνετε και ε, έργα, να μην περιοριστείτε στα λόγια όπως για την περίπτωση του κράτους δικαίου, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και όλων των πολιτών των δικαιωμάτων, δηλαδή και των προσφύγων και μεταναστών. Ευχαριστώ πολύ κυρία Ντέλη, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο Πρωθυπουργό είπε ότι μία προτεραιότητα είναι η διασφάλιση των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Κροατία όμως πώς μπορεί να καθοδηγήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ζητήματα βέλτισης πρακτικής όσον αφορά το άσυλο και τη μετανάστευση και ιδίως όσον αφορά τη σχετική τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όταν υπάρχουν τόσες τεκμηριωμένες πληροφορίες για τη χρησιμοποίηση αστυνομική βίας κατά των μεταναστών και την παράνομη επαναπροώθηση μεταναστών προς τη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Πρόκειται για πρόδειλη παραβίαση του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, καθώς επίσης και της Σύμβασης για τους Πρόσφυγες. Δύο Νιγηριανοί αθλητές μάλιστα συνελήφθησαν ανάμεσα στους υπόλοιπους μετανάστες στο Ζάγκρεμπ και πραγματικά συμμετέχοντας στην Ευρωπαϊκή Πολιτικών Ελευθεριών Διερωτώ με, είναι ποτέ δυνατόν να χρησιμοποιούμε εκατομμύρια ευρωπαϊκούς πόρους προκειμένου να έχουμε ένα μηχανισμό παρακολούθησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όταν βλέπουμε ότι ένα κράτο Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν παραβιάζει τους κανόνες αυτούς. Ο κύριος Μπόκοβιτς έχει το λόγο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρώην συνάδελφο Αντρέι Πλέκοβιτ Καλώ ε, ήρθε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Χαίρομαι πάρα πολύ που σε ξαναβλέπω εδώ και χαίρομαι πάρα πολύ που αναλαμβάνει την πρώτη αυτή Προεδρία του 2020 η Κροατία. Η Ευρώπη σίγουρα αντιμετωπίζει πολλέ διαφορετικέ προκλήσει. Εγώ με τη σειρά μου θα ήθελα να επικεντρωθώ στο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Ελπίζω ειλικρινά ότι ω ένα νέο κράτο μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, που γνωρίζετε πόσο σημαντικά είναι τα γεωργικά ταμεία και το Ταμείο Συνοχή, θα επικεντρωθείτε πάρα πολύ στο ζήτημα αυτό του πολιετέ δημοσιονομικού πλαισίου. Απότερο στόχο του, τελευταία ανάλυση, είναι να έχουμε μια ισότιμη ανάπτυξη σε όλε τι περιφέρειε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίση, είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να χειριστούμε καλύτερα τη μετανάστευση. Εγώ ασχολούμαι με ένα πρόγραμμα το οποίο έχει να κάνει με τα ευφύ χωριά και τι κομοπόλει. Θέλουμε να αυξήσουμε την ψηφιοποίηση των περιοχών αυτών και θέλουμε μέσω της ψηφιοποίησης να οδηγηθούμε σε καλύτερη οικονομική ανάπτυξη και περισσότερες θέσεις απασχόλησης. Ο κύριος Λόπες Αγγιλάρο, τελευταίος ομιλητής στα πλαίσια δικασίας Catch the Eye. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρωθυπουργέ Πλένκοβιτς, όντως είναι η πρώτη φορά που η Κροατία θα ασκήσει την Προεδρία, την εναλλασσόμενη Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ε, της ευχόμαστε τα καλύτερα και την χαιρετίζουμε. Ταυτόχρονα υπογραμμίζουμε ότι είναι μια ευκαιρία που δεν θα πρέπει να τη διασπαθήσετε. Να κάνετε τη διαφορά σε σχέση με, τα, με τις κακές προβλέψεις που προϊονίζεται το ΠΔΠ σε ό,τι αφορά την συνοχή και την περιφερειακή πολιτική γιατί ε, αυτή είναι η προτεραιότητα και απόλυτα συμβατή με, τον, με τη νέα πράσινη συμφωνία. Μπορούμε να διαφυλάξουμε και τις πολιτικέ. πολιτικές. Επίσης, θα ολοκληρωθεί το Brexit στη διάρκεια της Προεδρίας σας. Ε, θα είναι ε, μέλημά σας, ελπίζω, να διασφαλίσετε αμοιβαιότητα και να εγγυηθείτε τα δικαιώματα των πολιτών και να δώσουμε στον χώρο ασφάλειας και δικαιοσύνης ε, τη θέση που το αξίζει γιατί το Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να αυτοεξαιρέθηκε από πολλέ πολιτικέ. Στη μελλοντική μα όμω σχέση θα πρέπει να δούμε ποιο θα είναι ο ρόλο του Ηνωμένου Βασιλείου σε θέματα συνεργασία, ασφάλεια και προστασία των δεδομένων. Γιατί έγιναν σοβαρέ παραβιάσει ε, στην αρχή τη ε, υποβολή ε, και μετάδοση διάδοση δεδομένων, μετάδοση δεδομένων σε τρίτε χώρε. Επίση, και ο χώρος του Σέγγεν είναι σημαντικό θέμα και χώρες όπως η δική σας έχουν απόλυτο δικαίωμα να απολαμβάνουν την ελευθερία της ε, διακίνησης των ατόμων. Σας ευχαριστώ και ο λόγος στην κυρία Φόντερ Λάιν για να απαντήσει. Thank you, Mr. President. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα αναφερθώ στα τρία θέματα τα οποία μας απασχόλησαν περισσότερο. Το πρώτο είναι βεβαίω ο προπολογισμό, το ΠΔΠ, το δεύτερο είναι το Brexit, το τρίτο είναι τα Δυτικά Βαλκάνια. Πρώτον, λοιπόν, όσον αφορά τον ε, προπολογισμό. Κύριε Πρωθυπουργέ, είναι σημαντικό η Κροατική Προεδρία να πείσει το Συμβούλιο να τηρήσει τα επισημένα. Χρειάζεται ένα εξυγχρονισμό του προπολογισμού. Γιατί αυτό. Ο προπολογισμό που έχουμε τώρα συμφωνήθηκε το 2013. Θυμάστε το 2013. Ήταν όταν εντάχθηκε η Κροατία. Ο κόσμος ήταν εντελώς διαφορετικός. Δεν είχαμε ε, ιδέα περί της ύπαρξης του Ισλαμικού κράτους. Υπήρχε, αλλά δεν το ξέραμε. Δεν είχε υπάρξει η μεταναστευτική κρίση. Η Ρωσία δεν είχε προσαρτήσει την Κρυμαία και δεν είχε ξεκινήσει τον υβριδικό πόλεμο στην Ουκρανία. Δεν υπήρχε η κλιματική συμφωνία των Παρισίων. Δεν μιλούσαμε για ε, πέμπτη γενιά κινητή τηλεφωνία ή τεχνητή νοημοσύνη. Λοιπόν, από αυτά τα λίγα θέλω να σα δώσω να καταλάβετε ότι είναι τελείω διαφορετικό ο κόσμο και χρειαζόμαστε τελείω διαφορετικό προπολογισμό. Ένα μήνυμα λοιπόν από μένα και νομίζω ότι εδώ με στηρίζει το Κοινοβούλιο. Εάν το πλαφόν είναι χαμηλό, εάν είναι πολύ μικρός ο προϋπολογισμός. Ο μόνος, η μόνη διέξοδος είναι ήδη πόροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και υπάρχει μια ευκαιρία να γίνει αυτό με το σύστημα εμπορίας εκπομπών. Γιατί τα έσοδα του συστήματος αυτού θα αυξηθούν. Οπότε δεν αφαιρούμε τίποτα από τα κρατημέλη. Αντιθέτως θα έχουν περισσότερα. Αλλά μπορούμε να α, και στο ευρωπαϊκό επίπεδο τα σχετικά έσοδα για να υπηρετήσουμε το ευρωπαϊκό Green Deal. Δεύτερον, Brexit. Η Προεδρία έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή γιατί πρέπει να σημειωθεί τεράστια πρόοδος μέχρι το τέλος Προεδρίας σας. Μέχρι το καλοκαίρι. Και πρέπει να αποφασίσουμε λοιπόν, το Ηνωμένο Βασίλειο δηλαδή, να αποφασίσει πόσο κοντά ή πόσο μακριά θέλει να είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην ενιαία αγορά. Εν ολίγης. Δεν μπορούμε να έχουμε ελεύθερη μετακίνηση ε, για τους ανθρώπους αλλά να, ή να μην έχουμε για τους ανθρώπους αλλά να έχουμε για αγαθά και υπηρεσίες. Είτε για όλα αυτά, είτε για τίποτα. Δεν μπορούμε να έχουμε ίσους όρους ανταγωνισμού, αν υπάρχει τεράστια απόκληση στη φορολογία ή στη κοινωνικά, τα περιβαλλοντικά και τα σχετικά. Είναι λοιπόν μια επιλογή του Ηνωμένου Βασιλείου κατά πόσον θέλουν να συγκλίνουν ή να αποκλίνουν, αλλά αυτό είναι αποφασιστικό για το πόσο ε, θα έχουν πρόσβαση στην κοινή αγορά ή όχι. Όπως λέγει η οχι οπως λεει η παροιμια δεν γίνεται και την πίτα ολόκληρη και το σκύλο χορτάτο. Τέλος για τα Δυτικά Βαλκάνια. Θεωρώ για τα Δυτικά Βαλκάνια δεν επιτρέπεται να το υποτιμάμε. Είναι προς το στρατηγικό μας συμφέρον τα Δυτικά Βαλκάνια να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά σε εμάς. Δεν πρέπει να υποτιμούμε την ήδη ισχυρή παρουσία της Κίνας, της Ρωσίας, της Τουρκίας. Όλοι είναι εκεί με την πρόθεση να ε, τραβήξουν τις χώρες αυτές ε, προς το δικό τους το μέρος. Πρέπει λοιπόν να τις φέρουμε πιο κοντά σε εμάς, ε, έχοντας λοιπόν κατά νου την Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία. Ζήτησαν πολλά πράγματα. Η Βόρεια Μακεδονία άλλαξε το όνομά της για να έχει την δυνατότητα να ανοίξει τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις. Λοιπόν, θα πρέπει να εξυγχρονιστεί αφενό η διαδικασία ένταξη, αλλά να τηρήσουμε και αυτά τα οποία είχαν προσχεθεί στι δύο χώρες. Είναι προ το συμφέρον μας. Αυτά και εύχομαι καλή επιτυχία στην Προεδρία σας. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Τον λόγο τώρα έχει ο κύριος Πρωθυπουργός. Αντρέη, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ. Ντάβιτε. Κυρίες και κύριοι, αγαπητέ Πρόεδρε, καταρχήν σας ευχαριστώ για τις αντιδράσεις σας, τις πολλές προτάσεις και τις διαφορετικές απόψεις για τις προτεραιότητες της Κροατικής Προεδρίας. Σας ευχαριστώ επίσης για τις ιδέες που εκφράσατε, για το πώς πιστεύετε ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τους πιο δύσκολους πολιτικούς και νομοθετικούς φακέλους. Να πω δύο λόγια καταληκτικά για να προσπαθήσω συλλογικά να αγγίξω κάποια από τα θέματα που θίξατε. Καταρχήν, ποια είναι η φιλοσοφία της ε, πρώτης μας προεδρίας. Είμαστε κατά κάποιο τρόπο ένα μήνυμα και ένα σύμβολο, το είπα και στην αρχή. Μόνο 30 χρόνια δημοκρατίας, 28 έτη διεθνούς αναγνώρισης και 7 έτη που είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξακολουθούμε να προσπαθούμε να φτάσουμε αυτούς που είναι πιο αναπτυγμένοι όσοι ήταν από την αρχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όσοι μπήκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004 και το 2007. Ο κύριος Κράχ, νομίζω, ένας ευρωβουλευτής, ανέφερε τον ε, κύριο Τουσμαν, τον πρώτο πρόεδρο της Κροατίας και προσπάθησε να ερμηνεύσει το δόγμα του. Εγώ θα ήθελα να πω ότι ίσω να γνωρίζω κάπω καλύτερα ποια είναι η κληρονομιά του πρώτου πρόεδρου της Κροατίας και το τι ήθελε για την Κροατία όταν κερδίσαμε την ανεξαρτησία μας για το μέλλον και για την προοπτική της χώρας. Ε, αυτός ήταν ε, μάλιστα πριν από 30 χρόνια στις 30 ε, Μαΐου, στο πρώτο, στις 13 χρόνια συγγνώμη, που είπε ότι η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση είναι οδός που πρέπει να ακολουθήσουμε και τα αυτά που κάναμε τις τελευταίες τρεις δεκαετίες ήταν η εφαρμογή του στόχου αυτού. Ξέρουμε τι σημαίνει η εθνική κυριαρχία σε αντίθεση με οποιαδήποτε άλλη χώρα που είναι εδώ στο ημικύκλιο, τι σημαίνει να έχεις κατεχόμενα εδάφη, τι σημαίνει να έχεις πόλεμο στα εδάφη σου και πάνω από 60.000 νεκρούς στη χώρα σου. Στα τέλη του 20ου αιώνα. Έχουμε ζήσει αυτή την εμπειρία και ξέρουμε ότι η Ευρώπη είναι ένα οικοδόμημα ειρήνης, ανοικοδόμησης και συμφιλίωσης. Και έτσι αντιμετωπίζουμε σήμερα την πολιτική μας ευθύνη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να σημειωθεί. Δεύτερον, λάβαμε υπόψη το, στρατηγική, το στρατηγικό θεματολόγιο, το πρόγραμμα του Τρίου του το πρόγραμμα της Νέας Κομισιόν και το δικό μας πρόγραμμα. Όλα όσα θέσαμε προτεραιότητες είναι πολύ ρεαλιστικά. Και επομένως για κάποια από τα σημεία ξέρουμε ότι η κλιματική αλλαγή και ο στόχος της κλιματικής ουδετερότητας μέχρι το 2050 θα είναι η ατμομηχανή της οικονομικής μας ε, μετάβασης. Ε, θα ε, είναι για την οικονομία ό,τι σημαίνει τα ανθρώπινα δικαιώματα στην εξωτερική μας πολιτική. Και αυτό συζητήσαμε στο Ζάκρεπ την περασμένη εβδομάδα. Θα λάβουμε υπόψη το διαφορετική κατάσταση των βιομηχανιών μας, ε, την οικονομική μας ικανότητα, τη δημοσιονομική μας ικανότητα προκειμένου να οδεύσουμε προς την ίδια κατεύθυνση και να μην έχουμε αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις. Δεύτερον, για το φάκελο της μετανάστευσης που πολύ αναφέρατε, θα πω εκ νέου. Και αυτό το επαναλαμβάνω γνωρίζοντας πλήρως ότι πρέπει να αναλάβουμε ζωτική δράση τους επόμενους μήνες. Έχουμε τη διευθέτηση με την Τουρκία που κατάφερε να μειώσει τον αριθμό των παραμεταναστών στην οδό της Ανατολικής Μεσογείου και των Δυτικών Λυκανίων κατά 98% αν συγκρίνουμε με τα στοιχεία του 2015-2016. 2015-2016. Αυτός τους αριθμούς έχουμε τώρα σε σχέση με 5 έτη πριν, 2%. Πώς θα το αντιμετωπίσουμε αυτό από κοινού. Μιλάμε για το ότι η Frontex θα έχει 10.000 συνοριοφύλακες. Ίσως η χώρα μου έχει τους περισσότερους από οποιαδήποτε άλλη χώρα. 6.500 συνοριοφύλακες. Ακούω κάποιους ισχυρισμούς και δηλώσεις ε, στις εκθέσεις που διαβάζετε, στις φήμες που ακούτε. Ε, ότι σχεδόν ε, είναι έτοιμο να λεπιθεί. Όχι. Υπήρξε μάλιστα, όποτε υπήρξε ισχυρισμό, υπήρξε και έρευνα. Υπάρχει ισχυρή παρακολούθηση εντό αστυνομία για να αποτραπεί οποιαδήποτε παραβίαση ανθρωπινών δικαιωμάτων, οποιασδήποτε συμπεριφορά που είναι παράνομη και δεν σέβεται τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τι διεθνεί συμβάσει. Αλλά επαναλαμβάνω εκ νέου, σε αντίθεση με πολλά άλλα κράτη-μέλη, έχουμε πει ότι δεν θα ε, έχουμε σειρματοπλέγματα μεταξύ Κροατία και Βορζία Ενσεκοβίνη και ούτε θα χτίσουμε τύχη μεταξύ των κρατών που είναι φιλικά κράτη και θα ε, συνεχίσουμε τη φιλική μας συνεργασία. Και είπαμε ξεκάθαρα, δεν θα υψώσουμε τύχη μεταξύ μερών των συνόρων της Βοσνίας Ερζεγοβίνης, όπου ζουν Κροάτες ως πολίτες της Βοσνίας Ερζεγοβίνης και Κροάτες από την άλλη πλευρά των συνόρων. Αυτό δεν θα συμβεί. Αυτή είναι η πολιτική μας και την υποστηρίζουμε. Αλλά τι θέλουμε να κάνουμε από κοινού, να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα είτε στην πηγή είτε στο πρώτο σημείο εισόδου. Το σύνορο του κρατια Βοσνία Βοσνία-Ερτσεγοβίνη δεν είναι το πρώτο σημείο εισόδου των μεταναστευτικών ροών. Α είμαστε ξεκάθαροι. Αυτό είναι σημαντικό να το σημειώσουμε. Για τον προπολογισμό. Έχουμε πολλά που διακυβεύονται. Κατανοήσαμε τα μηνύματα ότι δεν μπορούμε να κάνουμε περισσότερα με λιγότερους σπόρους. Ξεκάθαρο είναι αυτό αλλά θα πρέπει να βρούμε μία συνένεση αν ε, θέλουμε να προχωρήσουμε προς τους νέους ίδιους πόρους. Είχαμε πολλές αναλύσεις ικανών ανθρώπων τα προηγούμενα έτη και από ό,τι φαίνεται αυτός είναι ο μόνος τρόπος, όπως είπε και η Ούρσουλα, να αντιμετωπίσουμε τις προσδοκίες ε, του εξυγχρονισμού για το τι μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε από κοινού. Αυτό είναι κλειδί, γιατί δημογραφικό αν υπάρχει ένα στοιχείο πολιτικό που θα ήθελα να φέρω ως κληρονομιά της Κροατίας και να αφήσω ως κληρονομιά της Κροατίας ε, το επόμενο εξάμεινο και έχει εκφραστεί αυτό, αυτό το χαρτοφυλάκιο για πρώτη φορά στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί θεωρούμε ότι είναι υπαρξιακό θέμα. Ε, γιατί τα μισά από τα κράτη-μέλη έχουν αρνητική ανάπτυξη, όπως και η δική μου χώρα. Νομίζω ότι να θέσουμε εργαλεία με την ευαισθησία της Προεδρίας της Κομισιόν, που ξέρει πόσο σημαντικός είναι αυτός ο ρόλος, να δούμε πώς μπορούμε να συνδυάσουμε μέτρα πολιτικής που έχουν αποδειχτεί αποτελεσματικά σε άλλες χώρες και πώς μπορούμε να τις προσφέρουμε τα μέτρα αυτά σε όσους έχουν δυσκολία. Αυτή είναι η ιδέα ο πληθυσμό ε, από λιγότερο αναπτυσσόμενε χώρε σε πιο αναπτυγμένε, από τι ε, αγροτικέ περιοχέ, τι αστικέ περιοχέ. Αυτά είναι κοινά προβλήματα που πρέπει από κοινού να αντιμετωπίσουμε. Για τα Δυτικά Βαλκάνια και το θέμα τη διεύρυνση. Δεν είμαστε αφελεί, ούτε μη ρεαλιστέ. Ίσως ε, ξέρω καλύτερα γιατί ασχολούμαι με αυτά τα θέματα για 30 χρόνια ότι το επίπεδο ενθουσιασμού απέναντι στην Δύση και το τι προσέφερε η Δύση τη δεκαετία του 90 στις χώρες της Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης δεν θα ξανασυμβεί σε αυτούς που θέλουν να προσχωρήσουν. Όμως πρέπει να έχουμε μια ευφυδομημένη προσέγγιση τα επόμενα δεκαέτη και να καθοδηγήσουμε αυτή τη διαδικασία, να προσφέρουμε φιλόδοξο θεματολόγιο για όσους θέλουν να κάνουν μεταρρυθμίσεις και να φτάσουν στα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή είναι η ιδέα πίσω από τη σύνοδο που θέλουμε να οργανώσουμε στο Ζάγκρεμ. Και επομένω λέω, για όσους φοβούνται να πούνε ναι στην ε, έναρξη της διαπραγματευτικής διάσκεψης με τη Βορεια Μακεδονία και την Αλβανία. Το ξέρουμε. Είναι μια διαδικασία πολύπλοκα, πολύπλοκη νομικά, με πολλές ε, δυνατότητες μπορεί να υπάρξει αναστολή, αναστροφή ή να ζητηθούν ακόμη περισσότερα όμως ε, πρόκειται για την αφετηρία ενός μαραθώνα. Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Δεν συμβαίνει εν μία νυχτή η διεύρυνση, συμβαίνει μετά από έτη πολλών ετών μεταρρυθμίσεων και προσεκτικού ελέγχου από την Κομισιόν και τη συνεισφορά των κρατών μελών. Δεν θα ήθελα λοιπόν καμία από τις χώρες στη γειτονία μας να ξεχαστεί, ιδίως η Βοσνία που είναι στρατηγική για τη χώρα μου. Επίσης, θέλω να αναφερθώ στην Ουκρανία, γιατί το αναφέρατε και εσείς τώρα, Ούρσουλα. Στο πλαίσιο της ανατολικής ε, γειτονίας ε, θα πρέπει να ε, δούμε ποιες είναι και οι δικές τους φιλοδοξίες για την εδαφική ακαιρεότητα αλλά και τις μεταρρυθμίσεις που πρέπει να υποστηρίξουμε για την ευρωπαϊκή προοπτική τους. Για τον Brexit βλέπω είναι εδώ Μισελ και αυτό το θέμα ακολουθεί τη συζήτηση. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό στοιχείο τα τελευταία 3,5 χρόνια ήταν η ενότητα των 27 χωρών. Παραμένουμε ενωμένοι, με πλήρη αλληλεγγύη, κυρίως για τις χώρες που τις αφορά περισσότερο όπως η Ιρλανδία. Το επόμενο ενδεκάμινο ε, θα, με, το, με ένα ε, πλαίσιο που θα το έχουμε διαπραγματευτεί και διατυπώσει καλά, νομίζω ότι μπορούμε να φτάσουμε σε ένα σημείο εφετηρίας για τη μελλοντική μας σχέση. Δεν θα ε, πρέπει ε, να θεωρούμε ότι μπορούμε να λύσουμε τα πάντα, το τι θα ισχύει στο μέλλον μετά το διαζύγιο που θα λάβει η χώρα σε τρεις εβδομάδες. Έτσι λοιπόν, βάσει της πρώτης κομισιόν θα εργαστούμε στο Συμβούλιο για να βρούμε την ορθή ισορροπία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας του επόμενου μήνες. Και τέλος να επαναλάβω ότι όλες μας οι υπηρεσίες, οι υπουργοί, η κυβέρνηση, οι ευρωβουλευτές που είναι εδώ και τους ευχαριστώ για τη συνεισφορά τους, θα είναι στη διάθεσή σας για να έχουμε έναν καλό διάλογο και να καταλήξουμε σε συμβιβασμού. Αυτό είναι από του στόχου τη Ευρωπαϊκή Δημοκρατία, αυτό είναι ο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κρατών μελών εντό του Συμβουλίου και επίσης ε, να διευκολύνουμε και τον ηγετικό ρόλο που έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρο για την ευκαιρία που μου δώσατε να σας απευθυνθώ εδώ σήμερα στο Στρασβούργο και μπορώ να πω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ένας πολύ αγαπητός θεσμός, ένα θεσμικό όργανο αγαπητό σε μένα. Ευχαριστούμε Πρωθυπουργέ Πλένκοβιτς, φυσικά να σας ευχηθώ κάθε επιτυχία στις εργασίες σας και κάθε επιτυχία στην κυβερνητική σας ομάδα για αυτή την πολύ σημαντική περίοδο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συζήτηση για το θέμα αυτό ολοκληρώνεται. Η διάταξη αναφέρει την διακήρυξη του Συμβουλίου και της Επιτροπής σε ε, σχέση με τις διατάξεις για τα δικαιώματα των πολιτών στη Συμφωνία Αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου. Παραμένει εδώ η πρόεδρος Φόντερ Λάιεν. Salutiamo e diamo la parola να δώσουμε το λόγο στην Υπουργό Εξωτερικών Νικολίνα Μπρνάτς, εξ του Συμβουλίου. Prego, λέει, la Έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη. Τώρα θα εξετάσουμε και μάλλον θα δούμε τη θέση σε ισχύ τη Συμφωνία Απόσυρση του Ηνωμένου Βασιλείου, που δεν έχει αλλάξει την ουσία από την προηγούμενη εκδοχή του 2019, εκτό από τι ε, διατάξει που αφορούν την Ελλαδία. Εμείς θέλαμε να μην αποδεχθούμε κάποια ε, άλλη ενθεώρηση των δικαιωμάτων των ε, πολιτών, όπως έχουν ζητήσει πολλοί. Γιατί αυτό θα έχει οδηγήσει σε μια αποδυνάμωση του επίπεδου προστασία από ό,τι έχουμε σήμερα, στο δεύτερο τμήμα της ε, συμφωνίας που έχει να κάνει με τα δικαιώματα των πολιτών. Κάτι το οποίο έχει ενταχθεί σε ολόκληρη τη συμφωνία και με συγκεκριμένες διατάξεις που προβλέπουν το ενδεχόμενο να μην υλοποιήσει ε, τα συμπεφωνημένα το Μνό Βασίλειο στο ακέραιο. Αυτό δεν σημαίνει ότι εμεί θα πρέπει να επαναπαυθούμε και είμαι ευγνώμων προ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που ε, έθεσε στην μισή διάταξη αυτό το ζήτημα σήμερα. Χαιρετίζω και το ψήφισμα που έχει κατατεθεί, γιατί αντιμετωπίζει ε, αρκετά από τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα δικαιώματα των πολιτών, τι διοικητικέ διαδικασίε που έχουν να κάνουν ακριβώς με αυτό το θέμα, την συνδρομή που παρέχει στους πολίτες και την αποτελεσματικότητα των ανεξάρτητων αρχών του Ηνωμένου Βασιλείου σε ό,τι αφορά την ε, ε, επίβλεψη και την εποπτεία των διαδικασιών αυτών. Αυτό δεν σημαίνει ότι και εμεί από πλευρά Ευρωπαϊκή Ένωση θα κάνουμε όλα τέλεια. Ε, είναι σημαντικό στο ψηφίσμα σα να σημειωθεί ότι θα πρέπει να ενθαρρυνθούν τα κράτη-μέλη να υιοθετήσουν καλύτερε διατάξει για το μέλλον των Βρετανών πολιτών που διαμένουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να επιμείνουμε ε, και από πλευρά ε, Ηνωμένων Βασιλικών, πλευρά Ευρωπαϊκή Ένωση οι ανεξάρτητε διοικητικέ αρχέ ε, να ασκήσουν τη δέουσα επιμέλεια σε ό,τι αφορά την υλοποίηση του δεύτερου τμήματο τη συμφωνία. Περισσότερα μένουν να γίνουν και σε ό,τι αφορά την επίγνωση των πολιτών και από τι δύο πλευρέ τη μάχη σε ό,τι αφορά τη συμφωνία απόσυρση και αποχώρηση. Ε, για τους πολίτες. Ε, είναι απαραίτητο, ιδίως για τους πλέον ευάλωτους, να ξέρουν ποιες είναι οι διαδικασίες και ποια είναι τα δικαιώματά τους. Και τα κοινοβούλιο σίγουρα μπορεί να διαρματίσει ρόλο σε ό,τι αφορά την ενημέρωση των πολιτών. Βέβαια, όλες αυτές οι διατάξεις ε, παρότι οι επιπτώσεις ε, θα ε, είναι σε ισχύ περισσότερο και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, δεν θα καλύπτει αυτούς που θα έρθουν στη συνέχεια. Παρότι γνωρίζουμε ότι η γραμμή της ε, κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου είναι να βάλει ένα τέλος στην ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η μελλοντική σχέση θα είναι φιλόδοξη και σε ό,τι αφορά την κινητικότητα. Αυτό θα πρέπει να συνοδεύεται και με την διατήρηση ορισμένων δικαιωμάτων των πολιτών. Κλείνοντα, θα ήθελα να σημειώσω το μεγάλο βαθμό σύγκληση που υπάρχει μεταξύ τη θέση σα ε, των ε, δικαιωμάτων των πολιτών, όπω έχει ε, σχεδιαγραφηθεί σε μια σειρά ψηφισμάτων και στι προτεραιότητε του Συμβουλίου. Αυτό δείχνει ότι έχουμε κοινού σκοπού ω τα δύο θεσμικά όργανα σε ό,τι αφορά το Brexit. Οι κοινέ μα προσπάθειε θα πρέπει να συμβάλλουν σε μια προσπάθεια διασφάλιση των δικαιωμάτων ε, των πολιτών κατά την ε, συμφωνία αποχώρηση, προκειμένου και οι Βρετανοί και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι υπήκοοι, αλλά και οι οικογένειέ του να συνεχίζουν να ζουν, να φοιτούν ε, ή να εργάζονται στη χώρα που έχουν επιλέξει. Ευχαριστώ πολύ την προσοχή σας. Να ακούσουμε τώρα την κυρία Φορντελάιν, την πρόεδρο Φορντελάιν. Έχετε το λόγο. you, Mr. Ε, ευχαριστώ, κύριε πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Την προηγούμενη εβδομάδα ήμουν στο Λονδίνο. Είχα την ευκαιρία να μιλήσω σε φοιτητέ ε, για την μελλοντική σχέση μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βεβαίως μεταδέχτηκα ερωτήσεις και η πρώτη ερώτηση που ακούστηκε ήταν δεν αφορούσε το εμπόριο, δεν αφορούσε τις οικονομικές υπηρεσίες, δεν αφορούσε την ασφάλεια, όσο σημαντικά και αν είναι αυτά τα θέματα, αφορούσε βεβαίως τα δικαιώματα των πολιτών. Και επανερχόταν η ίδια ερώτηση με διαφορετικές ε, ιστορίες. Ο ένας ήταν ένας νεαρός από το Μπενελούξ που ζούσε στο Λονδίνο. Μία άλλη ήταν μια Βρετανίδα κυρία με ε, Ιταλό σύζυγο και ανησυχούσε. Και οι ερωτήσεις ήταν ε, ελαφρώς διαφορετικές βεβαίως, αλλά οι λόγοι ήταν πάντα οι ίδιοι. Ο κόσμος θέλει ασφάλεια για την ζωή τους, για το μέλλον τους και για τους οικείους τους. Μιλάμε για 3,5 εκατομμύρια πολίτες στο Ηνωμένο Βασίλειο από τα κράτη-μέλη της Ένωσης και σχεδόν 1 εκατομμύριο Βρετανούς που ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μεγάλη αριθμή, αλλά πίσω από αυτούς τους αριθμούς κρύβονται άνθρωποι με την προσωπική τους ιστορία. Κάποιοι είναι πολίτες άλλης χώρας της Ένωσης που έχουν γεννηθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο, Άλλοι έφτασαν αργότερα. Πολλοί από αυτούς παντρεύτηκαν, έχουν παιδιά, πήγαν στο πανεπιστήμιο, ξεκίνησαν να δουλεύουν και εργάζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, διδάσκουν ε, παιδιά, νοσηλεύουν ασθενείς, ε, φροντίζουν τους γέρους. Ξεκίνησαν επιχειρήσεις και απασχολούν και άλλους ανθρώπους. Οπότε όποια και αν είναι η προσωπική τους ιστορία, έχουν ένα κοινό στοιχείο. Θέλουν ηρεμία. Θέλουν να μπορούν να προγραμματίσουν το μέλλον τους και το μέλλον των οικογενειών τους για να μπορούν να αισθάνονται στο σπίτι τους εκεί που βρίσκονται. Οπότε, κυρίε και κύριοι βουλευτές, η προστασία των δικαιωμάτων αυτών των πολιτών είναι η πρώτη μας προτεραιότητα από την στιγμή που βγήκε το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, χάρη στην εξαιρετική δουλειά του Μισελ Μπαρνιέ και της ομάδας του, η Συμφωνία Αποχώρησης παρέχει εκτεταμένες εγγύησεις για αυτούς τους πολίτες, τους δίνει την προστασία και την βεβαιότητα που χρειάζονται, τους επιτρέπει να παραμείνουν εκεί όπου βρίσκονται σήμερα, υπό τις ίδιες συνθήκες, για όσο επιθυμούν χωρίς καμία διακριτική μεταχείριση με βάση την υπηκότητα. Η συμφωνία αυτή και τα όσα έχουμε συμφωνήσει βεβαίως σημαίνει ότι έχει σαφείς υποχρεώσεις και το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ευρωπαϊκή Ένωση για να εγγυηθούν αυτά τα δικαιώματα. Είναι άλλο το να τα έχουμε σε ένα κομμάτι χαρτί και άλλο να ισχύσουν. Οπότε όταν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κυρώσει αυτή τη συμφωνία θα φροντίσουμε να την εφαρμόσουμε και το πνεύμα και το γράμμα της και βεβαίως πρόκειται για κάτι το ηθικό για εμένα. Υπάρχει εδώ μια ηθική επιταγή. Θα πρέπει να εφαρμόσει το σχετικό σχέδιο το Ηνωμένο Βασίλειο. Μέχρι στιγμής γύρω στα 2,5 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες έχουν ήδη ζητήσει ε, άδεια παραμονής. Οι περισσότεροι την έχουν ήδη λάβει και αυτό είναι κάτι πολύ θετικό. Αλλά γνωρίζετε ότι υπάρχουν περιπτώσεις ε, που έχουν απορριφθεί και ε, πολλοί ακόμα δεν έχουν κάνει έτσι. Υπάρχουν διάφορες ανησυχίες ε, που γύρονται οι γνωστές περιπτώσεις των, του Γάλλου Φούρναρη και του Πολωνού Σεφ. υπάρχουν και άλλες πολλές περιπτώσεις όπου ε, ο κόσμος δεν μπορεί να κάνει έτσι για οποιονδήποτε λόγο. Οι άλλοι έχουν λάβει, τους έχει ζητηθεί μάλλον, τους έχουν ζητηθεί περισσότερα αποδεικτικά στοιχεία παρά το ότι ζουν στη χώρα 14 χρόνια ας πούμε. Οπότε θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν αυτά τα ζητήματα, να μην υπάρχει καμία διακριτική μεταχείριση ή επιπλέον πολυπλοκότητα στην διαδικασία. Πρέπει να φροντίσουμε όλοι οι πολίτες, ειδικά οι πιο ευπαθείς, να υποστηριχθούν στην όλη αυτή η διαδικασία και πρέπει να φροντίσουμε η ανεξάρτητη αρχή παρακολούθησης να είναι ε, πλήρως ανεξάρτητη στην πραγματικότητα. Η Κομισιόν θα παρακολουθεί στενά την εφαρμογή. Είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε τους πολίτες της Ένωσης που ζουν στο Ενωμένο Βασίλειο για να έχουν την στήριξή μας και βεβαίως το ίδιο θα κάνουμε και για τους Βρετανούς πολίτες που ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα αυτά τα έχω θέσει και στον κύριο Πρωθυπουργό την προηγούμενη εβδομάδα όταν επισκέφθηκα το Λονδίνο. Θα συνεργαστούμε στενά με το Ηνωμένο Βασίλειο για να τα επιτύχουμε αυτά και να λύσουμε τα όποια προβλήματα το συντομότερο δυνατόν. Τέλος, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Τα καλά νέα είναι ότι θα υπάρξει συνέχεια ε, για τους ε, Ευρωπαίους πολίτες που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και αντιστρόφως ε, μετά το τέλος της μεταβατικής περίοδου αλλά μετά το τέλος της μεταβατικής περίοδου το Ηνωμένο Βασίλειο θα είναι τρίτη χώρα και το Brexit θα σημάνει άλλαγες για αυτούς οι οποίοι θα θελήσουν να συνεχίσουν να ζουν και στις δύο όχθες της μάχης. Θα πρέπει να διαπραγματευτούμε νέες σχέσεις και προετοιμαζόμαστε για την διαπραγματευτική εντολή για τις διαπραγματεύσεις αυτές πριν από την 1η Φεβρουαρίου. Όπως και στο παρελθόν και εδώ τα δικαιώματα των πολιτών θα είναι η πρώτη προτεραιότητα και θα διαπραγματευόμαστε πάντα καλόπιστα για να υπάρχει μια νέα ε, εταιρική σχέση με τους Βρετανούς φίλους μας. Όπως είπα και στους φοιτητέ εκεί στο Λονδίνο ε, είναι η γνωστή ιστορία για τους παλιούς φίλους που θα κάνουν μια νέα αρχή. Ευχαριστώ. Τώρα θα ακούσουμε τους εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων. Για το ΕΛΚ η κυρία Χιούμπνερ για τρία λεπτά. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, καθ' όλη τη διαδικασία του Brexit στο Κοινοβούλιο συναντηθήκαμε πολλάκι με τους πολίτες και με Βρετανούς πολίτες. Ακούσαμε ιστορίες και καταλάβαμε καλύτερα τις συνέπειες του Brexit για τα δικαιώματά τους ως Ευρωπαίοι πολίτες. Και οι ανησυχίες τους είναι και δικές μας. Σε όλα τα ψηφίσματα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναφέρθηκε στα θέματα των δικαιωμάτων των πολιτών, όμως τώρα υπάρχει το θέμα της βιωσιμότητας εξού και το νέο ψήφισμα. Η πλήρη εφαρμογή των νομικών λύσεων για τα δικαιώματα των πολιτών θα έχει μαζικό αντίκτυπο, ε, μεγάλο αντίκτυπο στη ζωή των πολιτών. Η εφαρμογή της Συμφωνίας Αποχώρησης έχει σημασία γιατί προσφέρει ελάχιστη ασφάλεια δικαίου στους ε, ανθρώπους. Έχουμε και το άρθρο 18, σημείο 4 της Συμφωνίας Αποχώρησης. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει αποφασίσει να υιοθετήσει την ε, προσέγγιση την ε, προσαρμογή για το πρόγραμμα της εγκατάστασης. Επίσης, λυπόμαστε που η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε την πρόθεσή της να θέσει τέλος στην ελεύθερη μετακίνηση των πολιτών στο μελλοντικό πλαίσιο συνεργασία. Οι Ευρωπαίοι πολίτε και οι Βρετανοί υπήκοοι έχουν αποφεληθεί ιδιαίτερα από την ελεύθερη μετακίνηση των πολιτών και ελπίζω να αλλάξει γνώμη η Βρετανική κυβέρνηση για αυτό το θέμα. Θα είναι επίση κρίσιμο να βρούμε τρόπου προ αμοιβαία αναγνώριση των προσόντων να είναι δυνατό για τους πολίτες να συμμετέχουν στις τοπικές εκλογές, να υπάρχει καλή συνεργασία στον τομέα του οικογενειακού δικαίου βάσει των διάφορων διατάξεων που υπάρχουν στο διεθνές δίκαιο και πιθανές αποκλήσεις ερμιστικές να μην θίξουν τα δικαιώματα των πολιτών. Εκτιμώ τις διασφαλίσεις που μας δόθηκαν από τη Βρετανική κυβέρνηση σε σχέση με τη λειτουργία της ανεξάρτητης αρχής παρακολούθησης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ωστόσο, θα παρακολουθεί την διαδικασία της εφαρμογής. Όπως τονίσαμε στο ψήφισμά μας, η μικρότερη μεταβατική περίοδος σημαίνει ότι θα έχουμε λιγότερο χρόνο για να θέσουμε σε εφαρμογή την διακυβέρνηση της ε, συμφωνίας για τα δικαιώματα των πολιτών ε, και μία εκστρατή ευαισθητοποίηση επίσης θα είναι προτεραιότητα. Τέλος, ε, η κατάλληλη και πλήρης εφαρμογή των δικαιωμάτων των πολιτών θα βοηθήσει να οικοδομηθεί η εμπιστοσύνη για τις επιτυχείς διαπραγματεύσεις για το μέλλον. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο κύριος Σίλβα Περέιρα για τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κύριε Μπαγνιέ, κύριοι συνάδελφοι. Βασικό μας ε, μέλημα εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και καθώς είμαστε μέλη που έχουμε εκλεγεί απευθείας από τους Ευρωπαίους πολίτες είναι να υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα όσων εκπροσωπούμε δημοκρατικά. Αυτό εξηγεί και γιατί βασική μας προτεραιότητα εδώ στο Brexit πάντα ήταν τα δικαιώματα των πολιτών. Όχι μόνο τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών που διαμένουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και τα δικαιώματα των Βρετανών πολιτών που διαμένουν σε όλη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε ακούσει ε, τις ε, σοβαρές ανησυχίες που έχουν εκφράσει τόσοι πολίτες και ΜΚΟ και έτσι δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το γεγονός ότι ο κόσμος πραγματικά ανησυχεί επειδή υπάρχει μεγάλος βαθμός αβεβαιότητας σε ό,τι αφορά τις ε, επιβλαβείς επιπτώσεις ε, του Brexit στη ζωή τους. Γι' αυτό βρισκόμαστε εδώ σήμερα, για να συζητήσουμε και να εγκρίνουμε ένα πολιτικό ψήφισμα που έχει κατατεθεί και χέρι τη στήριξη ε, πολλών πολιτικών ομάδων στο Κοινοβούλιο και έτσι να αποστείλουμε ένα ισχυρό πολιτικό μήνυμα. Η κυβέρνηση του Ερμηνού Βασιλείου μπορεί να κάνει περισσότερα και θα πρέπει να κάνει περισσότερα για να διασφαλίσει την πλήρη προστασία των ε, δικαιωμάτων των πολιτών στο πλαίσιο του Brexit. Σαφώς και αναγνωρίζουμε τις προσπάθειες που έχουν γίνει σε ένα τόσο δύσκολο ζήτημα. Όμως η αλήθεια είναι ότι η συμφωνία αποχώρησης ε, θα μπορούσε να είναι ακόμα πιο φιλική προς το χρήστη. και να υπάρχει ακόμα περισσότερη αρρωγή προς ε, τους πιο ηλικιωμένους και πιο ε, ευάλωτους πολίτες. Θα ήταν καλύτερο να διασφαλίσουμε την σωστή ε, αναθεώρηση της συμφωνίας από μια ανεξάρτητη αρχή. Επίσης, θέλουμε ένα κείμενο στα χέρια μας για να υπάρχει μεγαλύτερη πολιτική βεβαιότητα και ασφάλεια στο μέλλον, όχι μόνο για τους πολίτες, αλλά και για τους εργοδότες ε, ε, και τους ε, ιδιοκτήτες ακινήτων. Ελπίζουμε να έχουμε θετική ανταπόκριση από την Βρετανική κυβέρνηση ό,τι αφορά τα δικαιώματα των πολιτών. Ευχαριστώ. Ε, Ο κύριος Βερχόφστατ, για τρία λεπτά. Ευχαριστώ. Το πρώτο που θέλω να πω είναι να ευχαριστήσω την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κυρία Φόντερ Λάιαν, καθώς και τον Μισελ Μπαχνιέ για την συνεχή και αμέριστη στήριξή του προ τους ε, ε, πολίτε και τα δικαιώματά τους και ελπίζω το κοινοβούλιο μα ε, όταν ψηφίσει, νομίζω αύριο είναι η ψηφοφορία, να εγκριθεί το ψήφισμα με μια τεράστια πλειοψηφία που θα μας δώσει έτσι μια εντολή για να κάνουμε τις τελικές συζητήσεις με τις Βρετανικές Αρχές την Πέμπτη με έχει προσκαλέσει ο κύριος Μπάρκλεϊ, καθώς και ο νέος Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, ο κύριος Σπίντσερ. Είναι σημαντικό λοιπόν να λάβει ευρεία στήριξη το ψήφισμα για να έχουμε πιο ισχυρή εντολή την Πέμπτη και την Παρασκευή. Υπάρχουν ακόμα στοιχεία για προβληματισμού, συνάδελφοι, που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Αν δεν γίνει αυτό τώρα, μέχρι τα τέλη του μήνα, δεν θα τεθούν επιτάπητος πριν από τα τέλη της χρονιάς. Δεν μπορώ να φανταστώ το Κοινοβούλιο να συζητήσει και να εγκρίνει μία συμφωνία ελευθερών συναλλαγών χωρίς να επιληθούν τα προβλήματα και ανησυχίε των Ευρωπαίων και Βρετανών υπηκών σε ό,τι αφορά την ελευθερία κυκλοφορίας. Αυτά, αυτές οι ανησυχίες έχουν ήδη αναφερθεί από άλλους συναδέλφους. Πρώτον, η αυτόματη αναγνώριση των δικαιωμάτων των πολιτών. Έχουμε κυβέρνηση των συντηρητικών που πάντα λέει ότι θέλουμε λιγότερη γραφειοκρατία. Ε, εντάξει, λιγότερη γραφειοκρατία. Ο καλύτερο τρόπο να γίνει αυτό είναι η αυτόματη αναγνώριση. Να μην χρειάζεται. Να μην χρειάζονται όλε αυτέ τι διαδικασίε. Δεύτερον, να έχουμε ένα κείμενο στα χέρια μα. Γιατί είναι απαραίτητο αυτό. Λένε οι Βρετανοί, όχι δεν χρειάζεται, έχουμε mail. Ναι, αλλά φανταστείτε να πάει κάποιο ε, να επιστρέψει στην Ευρώπη και να πάει να ξαναγυρίσει στο Αρμίνο Βασίλειο και να του πούνε πού είναι τα εγγραφά σου. Α, δεν έχω. Έχω mail, αλλά έχω ξεχάσει το κινητό στο σπίτι, δεν έχω μπαταρία. Δεν μπορεί να μπει αυτό ο άνθρωπο ξανά στο Ηνωμένο Βασίλειο. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα έγγραφο στα χέρια μα. Αυτό είναι το δεύτερο στοιχείο. Και τρίτον είναι η ανεξάρτητη αρχή παρακολούθηση. Η πρότασή μου είναι απλή. Να έχουμε μερικού εκπροσώπους των τριών εκατομμυρίων. Και έτσι επιλύεται το πρόβλημα. Νομίζω θα πρέπει να εξετάσουμε αυτά τα ζητήματα και να τα επιλύσουμε εν ώψη της συνάντησης ε, την Πέμπτη και την Παρασκευή. Και Λίγη ευελιξία ζητώ μόνο από τον Πρωθυπουργό κ. Τζόνσον να πάρει και να ακολουθήσει το παράδειγμα τη Βασίλισσα ενδεχομένω. Γιατί χθε ε, δέχθηκε η Βασίλισσα να δώσει ε, μια ε, φάση μετάβαση προ τον πρίγκιπα Χάρη και έτσι μπορεί να κάνει το ίδιο και ο κ. Τζόνσον. Ευχαριστώ για τους πράσινους, ο κύριος Λαμπέρτς. Ευχαριστώ. Συχνά παρουσιάζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση ως ε, ένα τεράστιο, κυρίως οικονομικό πρόγραμμα που προωθεί τους κεφαλαίουχους. Υπάρχει αλήθεια εκεί, αλλά δεν είναι μόνο αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα 3 εκατομμύρια των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ζουν στον Ηνωμένο Βασιλείο και τα 2 εκατομμύρια Βρετανών που ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση το ξέρουν καλά. Η ελευθερή κυκλοφορία, η ελευθερία να εγκατασταθεί κανεί για να εργαστείς, να σπουδάσεις, ε, για να πάρεις τη εξίσου μια ελευθερία που παρέχεται σε όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωση. είναι πιθανότατα ένα από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ένωση και Ακριβώς ε, αυτό κινδυνεύουν να χάσουν οι πολίτες ε, με την ε, αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό το κοινοβούλιο και ο Μισελ Μπαρνιέ ασχοληθήκαμε να κάνουμε τα πάντα για να περιορίσουμε όσο δυνατόν περισσότερο τις ζημίες γιατί υπάρχουν ζημίες που προκαλούνται από την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύω ότι όσα τέθηκαν στη Συμφωνία αποχώρηση είναι ικανοποιητικά, αλλά έχουμε ένα πρόβλημα εμπιστοσύνη με το Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι αλήθεια ότι οι διοικητικές δυσκολίες ε, ε, υπάρχουν. Είναι αλήθεια ότι αυτή η απειλή ε, που έχει γραφτεί στο ε, Βρετανικό Δίκαιο Συμφωνία Αποχώρηση που προβλέπει δυνατότητα η Βρετανική κυβέρνηση να καταργήσει απλώ την ανεξάρτητη αρχή που θα παρακολουθεί την εφαρμογή τη Συμφωνία Αποχώρηση σε ό,τι αφορά το σεβασμό των δικαιωμάτων των πολιτών, όλα αυτά μα ανησυχούν. Επίση, οι διακήρυξει και δηλώσει κάποιων από το Υπουργείο Εξωτερικών που παρουσιάζουν ε, του πολίτες που κατοικούν στο Ευρωπαϊκό Βασίλειο ως απειλή για την ασφάλεια. Έτσι λοιπόν το μήνυμά μου στη Βρετανική κυβέρνηση είναι το αξί. Αν ε, πράγματι θεωρείτε την Ευρωπαϊκή Ένωση ως φιλική δύναμη στο Ηνωμένο Βασίλειο να δράσετε έτσι ώστε οι στάση σας, με τις στάσεις απέναντι στους Ευρωπαίους πολίτες να επιβεβαιώσετε αυτό το φιλικό καθεστώς, να μεταχειριστείτε του Ευρωπαίου πολίτε που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο όπως θα θέλετε θέλετε να μεταχειριστούμε εμείς τους Βρετανούς πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ. Για την ομάδα ID, ο κύριο Μπέκ. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι.